Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε τη Σύνοδο της Ολομελίας. κηρύσω την έναρξη της ε, Συνόδου η οποία διακόπτει την 11η Οκτωβρίου 2011. Τα πρακτικά της του 12 και 13 Οκτωβρίου είναι ήδη στην διάθεσή σας. Υπάρχουν παρατηρήσεις σχετικά με τα λογοπρακτικά. Όχι, θεωρούνται λοιπόν ως εγκεκριμένα. Θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Αυτή η εβδομάδα είναι πολύ σημαντική για την Ευρώπη. Χθες συμμετείχα στην συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Την Τετάρτη θα έχουμε την διάσκεψη του Eurogroup και το, θα έχουμε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα οποία συμμετέχουν ε, μέλη της ζώνης ευρώ και θα ληφθούν πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις για τις αγορές αλλά και για τους πολίτες μας. Ο κ. Βαν και ο κύριος Μπαρόζο θα βρεθούν ανάμεσά μας ε, την Πέμπτη όπου και θα έχουμε μια συζήτηση για την ε, κατάσταση. Αύριο έχουμε προβλέψει μια πολύ σημαντική συζήτηση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αλλά και ψηφοφορίε επί των προπολογισμού που προβλέπονται την Τρίτη. Επιθυμούμε ο προπολογισμό αυτό θα είναι ένα προπολογισμό για την ανάπτυξη, την ανάκαμψη και την αύξηση τη απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ όλου του συναδέλφου που έλαβαν μέρο στην διάσκεψη που ασχολήθηκε με το νέο πολιετέ ε, δημοσιονομικό πλαίσιο για το έτη 2014-2020. Σας υπενθυμίζω πως ε, πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς ε, λάβαμε την πρωτοβουλία αυτή για να διεξαχθεί η συζήτηση. Η συζήτηση αυτή πραγματικά εστέφθη από επιτυχία και προτείνουμε να συνεχιστεί η συζήτηση αυτή σε έξι μήνες, σε ένα χρόνο ακόμα θα ήθελα να τονίσω την συμμετοχή εκπροσώπων από τουλάχιστον 30 ευρωπαϊκά κοινοβούλια κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Το Ευρωκοινοβούλιο ε, συμμετείχε ιδιαίτερα έντονα στις συζητήσεις τώρα. Ε, η Τινήση, γνωρίζετε, χθες ε, για πρώτη φορά ψήφισαν σε ελεύθερες εκλογές. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για την Τινησία και για ολόκληρο τον αραβικό κόσμο οι εκλογές διεξήχθησαν ε, με ειρηνικό τρόπο, δεν υπήρξε βία. Ε, το ποσοστό συμμετοχής ήταν ιδιαίτερα υψηλό, έφτασε στο 90%. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην, προσεχή, στην κυβέρνηση. Μια αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν επιτόπου και σύντομα θα λάβουμε μια, την έκθεση αυτής της ε, ομάδας ε, παρακολούθησης ε, των εκλογών. Εγώ ε, στο προσεχές μέλλον θα μεταβώ στην την Ισία. Όλοι θεωρούμε ότι είναι ένας τόπος, ένας ιδιαίτερα σημαντικός για την Βόρειο Αφρική. Γνωρίζετε ότι η Βόρειο Αφρική παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη σχέση μας με την περιοχή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το νέο κοινοβούλιο θα πρέπει να στηριχθεί στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών, στον σεβασμό των ε, ελευθεριών. Θα μεταβώ το Σαββατοκύριακο στην Λιβύη να συζητήσω τα θέματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία, με ιδιαίτερη ικανοποίηση. μετά από στην χώρα αυτή, την ε, χώρα η οποία πλέον είναι ελεύθερη, διότι τα τελευταία 40 χρόνια, 40 χρόνια της δικτατορίας του Καντάφη υπέφερε η χώρα και ο λαός μαζί της. Τώρα, την περασμένη εβδομάδα λάβαμε μια πολύ σημαντική πληροφορία που εμφορά την Ισπανία και ολόκληρη την Ευρώπη. Η ΕΤΑ δήλωσε πως θα εγκαταλείψει τον ένοπλο αγώνα και αυτό πάει βήμα-βήμα με τη διάλυση της ε, χερχές με τη διάλυση της οργάνωσης ε, θα παραδώσουν τα όπλα τα μέλη της ε, ΕΤΑ με εκτιμάμε ιδιαίτερες προσπάθειες που κατέβαλαν οι Ισπανικές αρχές αλλά και όλες οι αρχές που αγωνίστηκαν κατά τη τρομοκρατία. Ήταν ένα μακροχρόνιο μια μακροχρόνια προσπάθεια και θέλαμε να χαιρετήσουμε τα οικογένειε των 829 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αυτής της 40 ετούς δράσης της ΕΤΑ τραγικές προφορίες ε, έφτασαν από την Τουρκία. Πάνω από 200 πρόσωπα έχασαν ε, την ζωή τους μετά από ε, τον σεισμό που έπληξε την χώρα. θα ήθελα εξ ονόματος του Κοινοβουλίου να εκφράσω τα συλληπιτήριά μας και την ελληνική στην οικογένειε των θυμάτων. Είμαστε στο πλευρό του τουρκικού λαού για την για το πλήγμα που υπέστη. Παρακαλώ, ενό λεπτού σιγή. Thank you. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτές ήταν οι ανακοινώσεις. Ε, τώρα, οι αρμόδιες αρχές της ε, Σουηδίας ε, μου ανακοίνωσαν την αναπλούση της κυρίας Λένα Εκ από τον κύριο Κεν Τζόχασον από την 18 Οκτωβρίου 2011. Καλωσορίζω τον νέο συνάδελφο.